Τέλος θα τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα σε μια ποιοτική υγεία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκροστέτ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η όλος παραδόξως κοινή συζήτηση για την όσο του Αλσχάιμερ αφενός και τους εισπνευστήρες για ασθματικούς αφετέρου. Θα ασχοληθούμε πρώτα με το τόσο σημαντικό αλλά και τραγικό θέμα που αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης κυρίας Ματίας με τίτλο «Την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την όσο του Αλσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας». Και μετά έχουμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους εισπνευστήρες για προφορική ερώτηση από την Επιτροπή Αναφορών. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ματίας για τέσσερα λεπτά, μια και είναι η εισηγήτρια τη έκθεση αυτή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη και πόσο επήγε αυτή η πρωτοβουλία. Αρχίσαμε πριν από έξι μήνες ε, το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ένα εξάμεινο πέρασε από την εκπόνηση της οδηγίας, από την έναρξη της εκπόνησης οδηγίας μέχρι την ψηφοφορία. Και σε αυτούς τους έξι μήνες πάνω από 700.000 άνθρωποι στην Ευρώπη ανέπτυξαν Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλη μορφή άνοιας. Και από μόνο το αυτό το αριθμητικό στοιχείο δείχνει πόσο επίγει η πρωτοβουλία αυτή, πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη της. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τους νοσούντες από αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας ε, είναι σημαντικές. έχουμε πάνω από 700.000 το χρόνο, πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη έχουμε να πάσχουν από άνοια ή Αλτσχάιμερ. Δεν μπορούμε φυσικά να κάνουμε διακριτική μεταχείριση μεταξύ των όσων ή μεταξύ των χωρών. Δεν μπορούμε να πούμε ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα πρέπει να δράσουμε σε πολλούς τομείς, σε πολλές διαστάσεις. Ε, η νόσος αυτή διπλασιάζεται κάθε, ο αριθμός των νοσούντων δρασουμε σε πολλους τομεις σε πολλες διαστασεις η νοσος αυτη διπλασιαζεται ο αριθμος των νοσουντων καθε 20 χρόνια. Αλλά ε, οι ρυθμοί αυτοί θα αυξηθούν στο μέλλον. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα, στην πρόληψη, να ανακαλύψουμε τι αιτίε αυτή τη νόσου. Γιατί είναι μια νόσος άγνωστη. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, περισσότερη συνεργασία, περισσότερους επιδημιολογικούς ελέγχους. Επίσης να δούμε πώς θα δώσουμε έμφαση στο θέμα της πρόληψης, να δούμε τους, τους παράγοντες κινδύνου. Χρειαζόμαστε ειδικευμένο προσωπικό. Θα πρέπει να καταρτήσουμε, να έχουμε πιο ειδικευμένους νοσηλευτές, να βοηθήσουμε τις οικογένειες, τους ασθενείς που έχουν δικαίωμα, που δικαιούνται αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να πατάξουμε τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και εντός ενός κράτους μέλους. θα πρέπει να έχουμε ε, ασθενείς πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα σχετικά με το φύλλο, με το τόπο κατοικία και με οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη από τις υπηρεσίες υγείας για τέτοιες νόσους. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και δεν μπορούμε ε, υπό το πρόσχημα της κρίσης να αγνοούμε αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικές και οι οικονομικές επιπτώσεις ε, τέτοιων ασθενειών. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να επενδύσουμε στους ανθρώπους, να επενδύσουμε στην πρόληψη, να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τους νοσηλευτές και τους παρέχοντες φροντίδες σε αυτούς τους ανθρώπους. Για κάθε ε, ασθενή από Αλσχάιμερ χρειάζονται τρεις που να το φροντίζουν. Ένας ε, ασθενής με Αλσχάιμερ δεν μπορεί να περάσει ούτε μια ώρα μόνος του χωρίς ε, παρακολούθηση χωρίς κάποιον να το φροντίζει. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε ανεξάρτητο καθένα στο δρόμο, το απομονωμένο, χωρί συνεργασία. Χρειαζόμαστε ελληνική για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτό το καυτό ζήτημα. Επίση, όταν μιλούμε για συνεργασία, όλοι γνωρίζουμε ότι κανεί δεν μπορεί απομονωμένα να επιτελέσει αξιόλογο έργο και να έχει θετικέ επιπτώσει. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλου του κοιόδη συγκητέ όλων των ε, πολιτικών ομάδων και να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν και στην ε, ομάδα μου, ιδιαίτερα τις γυναίκες που με βοήθησαν. Γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τα θέματα αυτά, είναι αυτές που φροντίζουν περισσότερο τους ασθενείς και ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα και πλήττονται και από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια συντονισμένη λύση για όλα αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς τον κύριο Επίτροπο. Τι προτάσεις, κύριε Επίτροπε, από αυτές που περιλαμβάνουμε στην έκθεση είστε διατεθειμένος να δεχτείτε και πότε ε, θα τις θέσετε σε ισχύ, γιατί πραγματικά, όπως είπαμε, είναι επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Ευχαριστώ για πέντε λεπτά. Το λόγο έχει η κυρία Ματσόνη που συνέταξε την προφορική ερώτηση για τους εισπνευστήρες, που είναι το δεύτερο σημείο της κοινής συζήτησης. Presidente, la ringrazio. Devo dire che eh, condivido anch'io. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ συμφωνώ ότι είναι περίπλοκη όλη αυτή η λογική διασύνδεση των δύο θεμάτων. Ε, όμως για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι σήμερα ασχολούμεθα με το θέμα αυτό. Ε, ένα θέμα το οποίο περιλαμβάνεται στην ερώτηση που υπέβαλα εκ μέρου της Επιτροπής Αναφορών. Αυτή λοιπόν η αναφορά αφορά την περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης στην Ευρώπη ε, που ε, της αρνήθηκε το δικαίωμα δικαίωμα ε, Αυτό παρουσιάστηκε και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ε, η υπόθεση λοιπόν αφορά ε, μια ιατρική συσκευή, συγκεκριμένα πρόκειται για έναν εισπνευστήρα για ασθηματικούς που είχε εμφανιστεί στην αγορά. Αυτό λοιπόν το προϊόν εμπιπτεί στην οδηγία την 9342 που προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια πιστοποίηση κατόπιν οι εθνικές αρχές είναι εκείνες που έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ε, τις ε, συσκευές αυτές. Ε, το προϊόν λοιπόν πουλήθηκε στην αγορά για πέντε χρόνια μέχρι το 96 με πολύ μεγάλη επιτυχία χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επιφύλαξη και μετά το προϊόν αυτό ελέγχθηκε από τις αρχές της Βαβαρίας η οποία ζήτησε από την Επιτροπή του Μαγδεμβούργου να αναθεωρήσει την άδεια που είχε χορηγήσει σε αυτή την επιχείρηση. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο ε, Υπουργός Υγείας της ε, Σαξονίας προχωράει στον έλεγχο και τελικά στο τέλος της διαδικασίας αναφέρει ότι οι πνευστήρες αυτοί ε, δεν είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές εκφράζει μάλιστα κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τις τις, ε, τα στοιχεία που ανέφερε η Βαβαρία και συνεχίζεται και αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνει ε, εξετάσεις και με βάση την ισχύουσα οδηγία. Την επόμενη τώρα χρονιά προέκυψαν ε, δραστηριότητες οι οποίες όμως δεν είναι τεκμηριωμένες. Εμείς ε, έχουμε λάβει υπόψη μας αυτές τις δραστηριότητες και το 1997 χωρίς να έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση στον ε, κατασκευαστή ο Υπουργός Υγείας, ο Ομοσπονδιακός αποφασίζει να αποσυρθεί το προϊόν από την αγορά. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει τέλος του 1997 είναι μια Οδηγεί που το άρθρο 8 ε, του 93-42. Εν τω όμως δεν υπάρχουν ε, καθόλου πληροφορίες. Δεν υπήρξε η φάση διαβούλευσης με τον κατασκευαστή. Γενικότερα λοιπόν επικράτησε μία σιγή και ο κατασκευαστής επειδή πίστευε ότι αυτή η σιγή σήμαινε κατ' ουσίαν την ε, απόσυρση των αμφιβολιών. Γι' αυτό ο κατασκευαστής επαναφέρει τη συσκευή αυτή το 2003. Δυστυχώς το 2005 και πάλι χωρίς καμία ιδιαίτερη ανακοίνωση οι γερμανικές αρχές αποφασίζουν εκ νέου ε, το προϊόν αυτό να αποσυρθεί από την αγορά. Πρέπει να διευκρινίσουμε ακόμα και σήμερα παρότι έχουν εκφραστεί πολλά αιτήματα, δεν έχει εμφανιστεί κανένα στοιχείο που να εξηγεί γιατί αποσύρθηκε αυτό το προϊόν. Άρα δεν υπήρξε ανακοίνωση, δεν υπήρξε άρνηση ε, οποιασδήποτε πραγματικότητας που να αφορά τον κατασκευαστή. Και υπήρξαν και πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τον κατασκευαστή, γιατί πάνω από 15 χρόνια περιμένει μία απάντηση και το προϊόν του δεν μπορεί να πωλείται στην αγορά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι και στα 6 χρόνια που πολύτο το προϊόν και επ' αυτού υπάρχουν στοιχεία τα οποία δόθηκαν και στην Επιτροπή σε αυτά τα έξι χρόνια εντωμεταξύ υπήρξαν ε, σημαντικές, ε, σημαντική εξοικονόμηση στις δημόσιες αρχές από ε, αυτό το προϊόν και υπήρξαν και πολλά, πολλές θετικές συνέπειες για όσους υποφέρουν από άσθμα. Ο κύριος Κλάιν, ο κατασκευαστής, αναφέρθηκε στην Επιτροπή Αναφορών η Επιτροπή ξεκίνησε την σχετική διαδικασία και για μεγάλο χρονικό διάστημα εξέτασε το θέμα αυτό το οποίο είχε σχέση με την αναφορά. Επίσης υπήρξε μια άτυπη διαβούλευση με τον Επίτροπο. Ζητήθηκε να δοθεί κάποια απάντηση διότι το αίτημα του αναφέροντος είναι ένα αίτημα το οποίο έχει σχέση με την επανεπιβεβαίωση της συμβατότητας του προϊόντος σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή εν να, δοθεί, να εκδοθεί μία απόφαση από το δικαστήριο. Όλα αυτά δεν συνέβησαν. Και κατά τη διάρκεια της συζήτηση που έλαβε χώρα στην Επιτροπή Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς ε, ε, δεν απάντησε για άλλη μια φορά στις ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή μας αποφάσισε, αποφάσισε το θέμα αυτό να το φέρει στην Ολομέλεια και εδώ να ζητήσει από την Επιτροπή σαφείς απαντήσεις. Διότι το θέμα αυτό ε, υπάρχει και προκαλεί πολλές και μεγάλες αμφιβολίες ω ως προς την παραβίαση του χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και όχι μόνο λόγω αδράνειας Επιτροπής αλλά και λόγω του ότι ε, ο κύριος Κλάιν, ο αναφέρον, δεν μπορεί να έχει μια δικαστική απόφαση. Η υπόθεση λοιπόν προκαλεί αμφιβολίες ε, όσον αφορά την ε, παραβίαση ε, των κανόνων της αγοράς και την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και εμείς να μας δοθούν κάποιες απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση που έχουμε καταθέσει. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ματσόνη και ευχαριστώ επίσης που εκφράσατε και εσείς την απορία σας και συμμερίζετε με ένα, τον προβληματισμό. Βεβαίω είναι πολύ σημαντική η ερώτηση, δεν αφαιρεί τη σημασία και εσείς ως πρόεδρος ε, της Επιτροπής Αναφορών θαυμάσια την παρουσιάσετε και είμαι μέλος της και εγώ και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον Επίτροπο και για τους βουλευτές τώρα να αναμίξουν δύο θέματα τόσο διαφορετικά μεταξύ του. φύση διαφορετικά. Και πραγματικά προβληματίζεται κανείς αν θα πρέπει να είναι κοινή η συζήτηση όπως ε, γράφει και στην ημερήσια διάταξη. Εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τζον Ντάλι, Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς επιτρέψτε μου να αποτίσω ένα φόρο τιμή στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην εισηγήτρια την κυρία Ματίας για την προσήλωσή της και τη δέσμευσή της στα θέματα αυτά του Αλτσχάιμερ και άλλων ε, ανιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως στους προβληματισμούς σας. Η άνοια σημαίνει μεγάλη οδύνη για εκατομμύρια Ευρωπαίων και των οικογενειών τους. Ε, με την ταχεία γύρανση του πληθυσμού τώρα έχει φτάσει η ώρα η Ευρώπη να δράσει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για την ε, Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες το 2009 για να βελτιωθεί η πρόγνωση, η διάγνωση, μάλλον η πρόληψη, η έρευνα και η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή η οποία συνεχίζεται και έχει παρουσιάσει και πάρα πολλές συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές και η έκθεση είναι πάρα πολύ επίκαιρες στη στιγμή που ε, τον ερχόμενο Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει σε κοινή δράση ε, Alcov ε, είναι η ε, ε, ονομασία αυτής της δράσης από τα αρχικά για την Αλτσχάιμερ και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Κοινή δράση λέγω που θα βασίζεται στην πρόληψη, το τονίζει και το Κοινοβούλιο στην εκθεσή του, αλλά και στη βελτίωση της γνώσης των στοιχείων και ε, στην ανταλλαγή των ε, πρακτικών. Και έναν άλλο τομέα θα αντιμετωπίσουμε που ζητάει το Κοινοβούλιο πραγματικά να δράσουμε. Τα δικαιώματα των ανθρώπων που νοσούν από την νόσο Αλτσχάιμερ Πραγματικά χρειάζεται συντονισμένη έρευνα για να δούμε πώς θα προλάβουμε ή θα καθυστερήσουμε την έναρξη της νόσου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των ευρωεκφυλιστικών νόσων, κυρίως ε, της Αλτσχάιμερ. Για πρώτη φορά 23 χώρες ε, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της Αλσάιμερ είναι καλή η πρόοδος που έχει γίνει στην Ευρώπη στη διάγνωση και στη θεραπεία και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προωθεί αυτό. Όπως συστήνει και το Κοινοβούλιο, στην πρωτοβουλία για τη στρατηγική της Ευρώπης το 2020 θα έχουμε κριτήρια για μια νέα εταιρική σχέση για την καινοτομία, ε, για μια γύρανση ενεργή και δραστήρια για να υποστηρίξουμε εδώ στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας ε, τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Και η πρωτοβουλία που λαμβάνεται για την υποστήριξη των ε, προσώπων που φροντίζουν ασθενείς με άνοιες και Αλτσχάιμερ. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βλέπει θετικά και άλλες συστάσεις του Κοινοβουλίου και μπορούμε να ε, ορίσουμε το 2014 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εγκεφάλου. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και τη Αλτσχάιμερ. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο της συζήτησης αυτής. Η αναφορά του κυρίου Κλάιν που είναι εφευρέτης και κατασκευαστής ε, του εφέκτο της συσκευής αυτής της πνευστικής. Η ε, κυκλοφορία του προϊόντος αυτού στην αφορά ε, η Γερμανία το 1997 δεν κατέστη δυνατή γιατί της το αρνήθηκαν. Δεν ε, δόθηκε συνέχεια ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε από τις γερμανικές αρχές, ούτε από τον κατασκευαστή τον ίδιο στην απόφαση αυτή. Στη συνέχεια, ο διανομέας είχε πει ότι θα έκανε και άλλες μελέτες πριν ξαναφέρει το προϊόν στην αγορά. Επανήλθε το προϊόν στην αγορά το 2002 με νέα ονομασία και πάλι απαγορεύτηκε από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές το 2005. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε μελέτησε προσεκτικά την περίπτωση και ολοκλήρωσε τη διαδικασία με μια επίσημη επιστολή στις γερμανικές αρχές και τον ίδιο το κατασκευαστή τον Ιούλιο του 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε ως εξή την κατάσταση. Η απαγόρευση από τις γερμανικές αρχές ήταν δικαιολογημένη διότι τα κλινικά στοιχεία που έδινε ο, κατα... κατασκευαστής ήταν ανεπαρκή για να αποδείξουν την ασφάλεια του ε, προϊόντος, τη συσκευή αυτή. Σύμφωνα με την οδηγία για τις ιατρικές συσκευέ, θα πρέπει να αποδεικνύει ο κατασκευαστή την ασφάλεια του προϊόντος για να μπορέσει να ε, χρησιμοποιηθεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά. Αυτό. Άρθρο 18 της οδηγίας ήταν εκείνο που βρήκε εφαρμογή που έχει να κάνει με περιπτώσει όταν κυκλοφορεί στην αγορά ε, ένα προϊόν ε, που φέρει την ένδειξη CE. Ε, στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε επίσημη απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν νομίζουμε ότι εφαρμόζεται εδώ διαδικασία ασφαλιστικής ρήτρας, γι' αυτό δεν χρειάζεται να ζητήσουμε ε, κοινοποίηση της απαγόρευσης του 2005 των γερμανικών αρχών. Τα εμπόδια που έχει τώρα ο κατασκευαστής να φέρει το προϊόν του στην αγορά είναι η απόφαση των γερμανικών αρχών του 2005. Η απαγόρευση. Δεν είναι απόφαση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, αναφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει ένδικα μέσα, ε, θα μπορούσε να το είχε κάνει σε εθνικό επίπεδο. Και όντως ε, έκανε χρήση αυτής της ευκαιρίας, αλλά οι ισχυρισμοί του απερίφθησαν από τα γερμανικά δικαστήρια. Θα ήθελα εδώ να τονίσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 κάλεσε τον αναφερόμενο να φέρει τη συσκευή ε, σε συμμόρφωση ε, με τις ισχύους διατάξεις, να φέρει τα κλινικά στοιχεία που ε, λείπουν για να συμφωνήσει με τις γερμανικές αρχές. Εξ όσων γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ίδιος αναφερόμενος δεν έδωσε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα ακούσουμε τώρα τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα, για δύο λεπτά, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το λόγο έχει η κυρία Ελένα Αντωνέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην όσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ματία στην εισηγήτριά μας για το έργο της. Εγώ ως και η εισηγήτρια του ΕΛΚ για το θέμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της έκθεσης. Η προσοχή και το ζωηρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το θέμα αυτό δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. 9,9 εκατομμύρια υποφέρουν από άνοια και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, αυτού του αριθμού αφορά πάσχοντες από Αλτσχάιμερ. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί ασθενεί που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί. Υπάρχουν ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την πρόσβαση στη θεραπεία και τη φροντίδα. Είναι κατακαιρματισμένε οι δράσει και άνισε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τέτοιου είδους νόσων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της εισπύρεσης των προσπαθειών για να καταπολεμήσουμε αυτή την νόσο και να προσθέσουμε μια νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και συντονισμένα μέτρα για να καταπολεμήσουμε προβλήματα που είναι κοινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υποστηρίζουμε την έκθεση την ελληνική μεταξύ των κρατών μελών και την ε, ανταλλαγή βέλτιστων προ... Ε, πρακτικών προκειμένου να αποφύγουμε επικάλυψη και κατασπατάληση πόρων. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της πρόληψης και η πρόορη διάγνωση στα αρχικά στάδια της νόσου. Αυτό είναι το κλειδί για να σημειώσουμε πρόοδο στην ε, καταπολέμηση αυτής της νόσου. Επίσης υπάρχει σχέση μεταξύ νευρολογίας και δημόσιας υγείας. Έτσι θα αποφύγουμε προβλήματα στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τα τεχνογνωσίας και την ε, αξιοποίηση της τεχνολογίας στην πράξη. Χρειαζόμαστε τέτοια πολυδιάστατη προσέγγιση για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη τη τεχνογνωσία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντωνέσκου. Εκ μέρους των σοσιαλιστών, το λόγο κυρία Childers για δύο λεπτά. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περίπου 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν σήμερα από άνοια και το Alzheimer είναι η πιο συνηθισμένη μορφή άνοιας. Η ίδια μου η μητέρα πέθανε πέρυσι από Alzheimer. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την άνοια. Ε, πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι μόνο το ίμιση των περιπτώσεων ε, είναι αντικείμενο διάγνωσης ε, και οι γυναίκες κυρίως διπλάσιος αριθμό των γυναικών που υποφέρουν από άνοια σε σχέση με τους άνδρες και πρέπει να ανησυχεί το ότι επειδή γυράσκει ο ε, πληθυσμό στην Ευρώπη θα διπλασιαστεί ο ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Ε, επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση πέντε ετών μέχρι να διαγνωστεί ασθένεια, εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προβάλλει ιδιαίτερα ε, την έγκαιρη διάγνωση. Καλύτερε έρευνε να υπάρξουν, κυρίω επειδή γνωρίζουμε ότι 85% των ερευνών σήμερα γίνονται χωρί να υπάρχει ευρωπαϊκό συντονισμό. Επίση, ε, χαίρομαι ε, και στηρίζω την διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Εγώ και οι σοσιαλδημοκράτε συνάδελφοί μου μου ε, ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα για την άνοια και λέμε το εξή. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στι ανάγκε των γυναικών, γιατί είπαμε ότι είναι διπλάσιο ο ρυθμό του ε, σε σχέση με του άντρε. Να την χάνουν σωστή θεραπεία, ε, η έρευνα μπορεί να βοηθήσει, όπω και σωστέ κοινωνικέ πολιτικέ. Καλούμε την Επιτροπή να νομοθετήσει για την πνευματική υγεία. Είναι δική τη η ευθύνη και η Επιτροπή πρέπει να εντάσει και στην αγορά εργασία άτομα με νευρικές διαταραχές. Υπάρχουν ε, επίσης ε, περιπτώσεις ε, στα σύνορα που έχουν ιδιαίτερε ανάγκες. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν και εκστρατείες για να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα συμπτώματα της άνοιας. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, την Μαρία Ματίας, να ευχαριστήσω τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, τους συναδέλφους μου για τη δουλειά που κάναμε όλοι για αυτή την έκθεση. Εκ μέρους των Φιλελευθέρων για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Φρεντερίκ Ρίς. Ευχαριστώ. Η καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ έχει γίνει μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι για τις πρωτοβουλίες που εξήγηλε ο Επίτροπος Ντάλι γιατί αυτή η μορφή εγκεφαλικής γύρανσης σοβεί 10 εκατομμύρια είναι περίπου οι άρρωστοι ε, από τέτοιε νόσου και από άλλε νευροεκφυλιστικέ νόσου και χαιρόμαστε για την ε, χρηματοδότηση 34 ερευνητικών σχεδίων με το θέμα αυτό αλλά θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι να βελτιώσουμε την προσπάθειά μα ιδιαίτερα στον τονισμό τη έρευνα ε, για το Alzheimer στα πλαίσια του 8ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου που πάει μέχρι το 2014. Αυτό αναφέρει το σημείο 21 του ψηφίσματος. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε μια πολυδιάστατη προσπάθεια που θα αφορά τη διάγνωση, την πρόληψη και την παροχή βοήθειας στους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους, το σημείο 20. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία μελέτη στη Γαλλία που ε, επισημαίνει ότι πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα είναι το κοινωνικό οικονομικό κόστος ε, της ε, φροντίδας ενός τέτοιου ασθενούς, χωρίς να υπολογίζουμε την αφοσίωση, την προσήλωση και το χρόνο που αφιερώνουν τα μέρη της οικογένειας έξι, έξι ώρες τη μέρα για την φροντίδα ενός τέτοιου ασθενούς. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε σφάλματα στη διάγνωση, γιατί μα το επισημαίνει ο επιστημονικό κόσμο. Θα πρέπει να τροποποιηθούν τα διεθνή κριτήρια. Γιατί εφαρμόζοντα κατά γράμμα κάποια παροχημένα κριτήρια, περιλαμβάνουμε πολλού ε, στην νόσο Αλτσχάιμερ ασθενεί που κανονικά νοσούν από άλλε νευροεκφυλιστικέ νόσου. Το σημείο 64 του ψηφίσματο είναι επίση σημαντικό και θα πρέπει να ακούσουμε την έκκληση των ερευνητών. Χρειαζόμαστε περισσότερου εθελοντέ ε, στι κλινικέ δοκιμέ για να βρούμε καλύτερες θεραπείες, γιατί η, η αναμενόμενη θεώρηση της οδηγίας είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανταποκριθούμε εμπράκτος στις ελπίδες αλλά και στις ανάγκες των οικογενειών των πασχόντων από Αλσχάιμερ. Εκ μέρους των Πρασίνων και για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Χέφνερ. Ja, wer immer das äh, veranlasst hat, diese Debatten zu Όποιος και αν είπε να συνδυαστούν αυτές οι δύο εισηγήσεις ε, δεν το σκέφτηκε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται το κόστος ε, των ασφαλιστικών ταμείων για θεραπείες ε, και πρέπει να δούμε πώς θα το μειώσουμε. Οι θεραπείες είναι όλο και πιο ακριβές. Εδώ όμως την περίπτωση που έχουμε, έχουμε να κάνουμε ακριβώς με το αντίθετο. Έχουμε 30 εκατομμύρια ασθματικούς ε, στην Ευρώπη και έχουμε έναν κύριο ο οποίος ε, έφτιαξε μια συσκευή με την οποία οι ασθενείς μπορούν να ζουν καλύτερα και μάλιστα και η θεραπεία τους είναι πολύ πιο προσιτή. Εδώ και 40 14 χρόνια με συγχωρείτε, ε, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να ε, παρουσιάσει και να ε, τοποθετήσει το προϊόν του στην αγορά. Η Επιτροπή Αναφορών επίσης ασχολείται με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν καθήκον της Επιτροπής, ε, κύριε Επίτροπε, να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να βρει το δίκιο του και να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τουναντίον η Επιτροπή αρνείται να λάβει μια απόφαση που θα βοηθήσει τον αναφέροντα και απευθύνομαι προσωπικά σε εσά κύριε Νταλή γιατί θα θυμάστε ότι σας καλέσαμε στην Επιτροπή Αναφορών για να συζητήσετε μαζί μας και μας είπατε δεν έχετε χρόνο, όμως είχατε χρόνο για προσωπική συζήτηση και ήρθαμε για προσωπική συζήτηση και εμένα προσωπικά μου υποσχεθήκατε ότι θα επιληφθείτε του θέματος και θα φροντίσετε ταχύτητα για μια λύση. Δεν άκουσα τίποτα μέχρι σήμερα. Σας έστειλα και επιστολή. Δεν απαντήσατε. Επίσης προσπαθήσατε να εμποδίσετε και την επόμενη συζήτηση. Ε, δεν πρέπει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν. Θέλω να πω, να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο περιμένει και αύριο θα ψηφίσουμε όλοι για αυτό το ψήφισμα. Περιμένει λοιπόν ο κόσμος, η Επιτροπή να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και ε, περιμένουμε από εσά ε, να προστατεύσετε αυτούς τους ε, μικρούς κατασκευαστές. Πρόκειται για πολλά χρήματα, πρόκειται όμως κυρίως για την υγεία των ανθρώπων. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και δεν κατανοούμε τις πράξεις σας κύριε Νταλή. Γνωρίζουμε τα επιχειρήματά σας. Διάβασα όλους τους φακέλους και δεν βρήκα κανένα πιστικό επιχείρημα που να ενισχύει τη θέση σας. Πρόκειται για μια ιατρική συσκευή. Έχει χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους με τα βέλτιστα αποτελέσματα και έχουμε επιστολές από ασφαλιστικές εταιρείε που ζητούν να επιτραπεί η χρήση αυτού του προϊόντος για να μειωθεί και το κόστος. Ε, παρακαλώ λοιπόν επιτέλους η Κομισιόν να καταλήξει μια θετική απόφαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάρτμουθ ε, έχει ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Κύριε Χέφνερ, το δέχεστε. Ο κύριος Ντάρτμουθ επιθυμεί να σας κάνει ερώτηση. Με γαλάζια κάρτα. Δέχεστε για 32 δεύτερα. Παρακαλώ. Μπορείτε να κάνετε την ερώτησή σας κύριε Ντάρτμουθ. Ντάρθμουθ. δεύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ θα συμφωνήσει μαζί μου ότι τα σχόλια του Επιτρόπου για το θέμα αυτό ήταν ε, πάρα πολύ ε, αόριστα, καθόλου χρήσιμα και για τους ε, ασθηματικούς αλλά και για τον κατασκευαστή της συσκευής αυτής. 30 δεύτερα. Επιτρέψτε μου να είμαι σύντομος και προσωπική είναι η απάντηση. Έχω την εντύπωση ότι ο Επίτροπος ακόμα δεν είχε την ευκαιρία να ε, ε, δημιουργήσει, να έχει τη δική του ε, άποψη. Όμως, κύριε Επίτροπε, προτείνω να καταφύγετε σε άλλους ε, συνεργάτες σας, ε, άλλοι και όχι παλιοί να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε εικόνα. Ε, θα ήθελα να το ξανασυζητήσω το θέμα μαζί σας. Βέβαια καλύτερα να καθίσετε με τον κατασκευαστή και να βρείτε μια λύση. Συμφωνώ απόλυτα, διακόπτει ο πρόεδρος τον κύριο Χέφνερ και του λέει τέλειωσε ο χρόνος σας. Τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γιανακουδάκη παρακαλώ εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. 750.000 ε, Βρετανοί πάσχουν από άνοια. Πάνω από τους μισούς έχουν Αλτσχάιμερ η εμπειρία του καθενό είναι διαφορετική, όσο ίδια και τα συμπτώματα. Χωρί θεραπεία είναι ανίατη η νόσου. Ε, όμοιροι είναι και ε, οι ασθενεί και εκείνοι που του φροντίζουν, ανεξαρτήτω ηλικία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η νομοθεσία είναι δευτερεύουσα. Αυτό που χρειάζεται κυρίω είναι επιτόπου υποστήριξη. Πρώτον, ε, να συζητηθεί αυτό το θέμα δημόσια και το πρώτο βήμα είναι στο Κοινοβούλιο. Ε, δημόσια συζήτηση, συνειδητοποίηση του κοινού για να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να το κάνουν προτεραιότητα και να μοιραστούν τις πρακτικές τους. Επίσης, η συνειδητοποίηση μπορεί να οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των συμπτωμάτων και συνεπώ σε έγκαιρη διάγνωση μπορούν να βοηθήσουν ενδιαφερόμενοι και εάν ε, εγκαίρως γίνει η διάγνωση μπορεί να επιβραδυνθεί η διαδικασία. Έτσι θα βοηθηθούν οι ασθενείς και οι οικογένειες και τελικά θα διασφαλίσουν και θα διατηρήσουν και την αξιοπρέπειά τους οι ασθενείς σε αυτή τη δύσκολη ασθένεια. Ευχαριστώ κυρία Γιανακουδάκη. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ντάτμουθ αλλά εξ ονόματος της ομάδας του, της Ευρώπης της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται, μια μικρή γερμανική εταιρεία Bronco Air του Μονάχου έχει φτιάξει μια συσκευή εισπνοής που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ασθηματικών που ε, ε, για να αναπνεύσουν ε, είναι εξαρτώμενοι από τέτοιες συσκευές. Πάνω από 14 χρόνια έχει αποκλειστεί από την αγορά αυτό το προϊόν. Και η εξήγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι συνέβη ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη τη Προέδρου τη Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή νομικών υποθέσεων είπε και παραθέτω ότι είναι θύμα κατάφορης άρνησης δικαιοσύνης η εταιρεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος παράθεσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευνοεί ε, τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και τα λόμπι. Το κόμμα μου, το κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ, ζητεί άμεση έρευνα στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ ο γύρος αυτός με την τοποθέτηση της κυρίας Ντότς, μισή λεπτό, εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων συναδέλφων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε ήδη σήμερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 750.000 ε, άνθρωποι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από κάποια μορφή άνοιας. Ε, 60.000 εξ αυτών ζουν την Βόρεια Ιρλανδία. Το Αλτσχάιμερ είναι μια φρικτή ασθένεια γιατί ε, σου αφαιρεί την ανεξαρτησία σου ε, και τελικά σου διαταράσκει τη σχέση σου με την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Πρόκειται για μια εκφυλιστική ασθένεια που ε, φέρνει μεγάλο βάρος για τις οικογένειες και τους νοσηλευτές. Οι άνθρωποι που φέρουν είναι απομονωμένοι και όπως αναφέρθηκε πολλοί από αυτούς που φροντίζουν ασθενείς είναι γυναίκες. Στο Ηνωμένο μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα υποφέρουν από άνοια θα εκτιναχθεί σε 1,7 εκατομμύρια και το προβλεπόμενο κόστος θεραπείας ε, θα ανέρχεται, ε, θα είναι υπέρογκο κόστος. Ε, μιλάμε για αριθμούς εντυπωσιακούς οι οποίοι καθιστούν απόλυτα απαραίτητη την έρευνα. Η πόροι πρέπει να χορηγούνται στοχευμένα στην θεραπεία. Ε, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη συνεισφορά των εθελοντών. Κύριε Επίτροπε, ε, μιλήσατε για τη γύρανση του πληθυσμού και εγώ είμαι περήφανη ε, που μπορώ να σας παρουσιάσω στο Belfast ένα πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει την απονομή βραβείων για εκείνους ε, οι οποίοι ε, φροντίζουν τους ανθρώπους που ζουν με άνοια και ζουν στις οικογένειές τους. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στους λοιπούς ομιλητές. Για 1,5 λεπτό πρώτα, ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε και εγώ το βρίσκω εκνευριστικό το ότι έχουμε τώρα να κάνουμε εδώ ε, με δύο θέματα, πάμε από το ένα στο άλλο. Εγώ θα ήθελα τουλάχιστον τα θέματα να εξετάσουμε το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, εγώ αναφέρομαι στην αναφορά του κυρίου Κλάιν και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό γιατί η Επιτροπή Αναφορών ασχολείται με το θέμα εδώ και αρκετό καιρό. Τι συνέβη ακριβώ. Υπήρξε ε, μια ε, καινοτόμα επιχείρηση η οποία κατασκεύασε έναν εισπνευστήρα για του ασθενεί ε, πολύ καλό για αυτούς ε, και για τα ασφαλιστικά ταμεία ε, και πολύ σωστά ο επιχειρηματίας βραβεύτηκε. Όμως μετά έρθε το σοκ. Οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν αυτό τον εισπνευστήρα. Γι' αυτό λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία ρήτρα διασφάλισης. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στην πρώτη απαγόρευση το 1996 δεν έγιναν όλα νομότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν υποχρεωμένη αυτή τη διαδικασία διαδικασία ρήτρα διασφάλιση, να την ολοκληρώσει με αποτέλεσμα ε, και να δώσει δυνατότητα στον ενάγοντα να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα. Ε, εδώ θα ήθελα να ε, παραθέσω τη θέση τη δική μα τη νομική επιτροπή. Σε τελική ανάλυση, ο κύριο Κλάιν είναι θύμα μια κατάφορη παραβίαση. Κύριε Επίτροπε, εμένα με ενδιαφέρει η απόδοση ευθυνών. Σημαντικότερο για μένα είναι να βρούμε το ταχύτερο δυνατόν μια λύση έτσι ώστε επιτέλους να αρθεί το πρόβλημα και σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας και την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής μας των Αναφορών. Εγώ λοιπόν εκ μέρους των αναφερομένων αλλά και εκ μέρους ε, των ε, ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να υπολογίζω ε, το πνεύμα συνεργασίας που θα επιδείξετε. Για 1,5 λεπτό η κυρία Σάρμπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ακόμη πολλές ε, αβεβαιότητες ό,τι αφορά τους ασθενείς ε, Alzheimer και δυστυχώς η κατάσταση θα επιδεινώνεται με την όλο και μεγαλύτερη γύραση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και περισσότερες μελέτες για τα αίτια και τη θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση ε, μορφών άνοιας. Μερικές φορές ακόμη και απλές αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης μπορούν να μας βοηθήσουν στην πρόληψη ε, τέτοιων ασθενειών, όπως ισχύει και για άλλες νόσους. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα διατροφής ε, ως μέσο πρόληψης της νόσου Αλσχάιμερ. Πολλοί από εμά γνωρίζουμε τουλάχιστον έναν ε, πάσχοντα, είτε από Αλσχάιμερ είτε από άλλη μορφή άνοιας. Και γνωρίζουμε ότι το προσωπικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο από το κοινωνικό ή το οικονομικό. Η άνοια, οποιαδήποτε μορφή άνοια, έχει καταστροφικά αποτελέσματα και αυτό είναι ανησυχητικό για όλους μας. Εξού και η έκθεση της κυρίας Ματίας που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Περιμένουμε θετική ανταπόκριση όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει η κυρία Παραβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τη δυσφορία μου για αυτή την κοινή συζήτηση ε, για δύο άσχετα θέματα. Είναι σαν να μιλούμε ταυτόχρονα για τα ναυπηγεία και την αλία μόνο και μόνο επειδή έχουν κοινό στοιχείο το νερό, το θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν έχουν καμία σχέση τα δύο θέματα μεταξύ τους. Πάντως χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ω προτεραιότητα την καταπολέμηση τη Αλσχάιμερ και άλλων μορφών άνοια. Είναι τεράστιο το βάρος των ε, συστημάτων υγεία μας από τέτοιες ε, νόσους, γιατί όχι μόνο αυτές οι νόσοι, αλλά και άλλες χρόνιες παθήσεις ε, θα αυξηθούν όσο γυράσκει ο πληθυσμός μας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρωτοστατήσει σε, στην πρωτοβουλία για τον Αλτσχάιμερ και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε δημόσιας υγείας εξαιτία του γυράσκοντα πληθυσμού χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη προσέγγιση και να επικεντρωθούμε στην έρευνα αλλά και στις στοχοθετημένες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Δεν θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε μόνο τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά να έχουμε κατά νου τη δημόσια υγεία και το συμφέρον των πολιτών. Γινόμαστε εδώ μάρτυρες ενός ε, λόμπι και των προσπαθειών ε, της ε, γερμανικής τοπικής αρχής να ευνοήσει τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε βάρο μιας μικρής. Αυτό που με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα για μα είναι το συμφέρον του καταναλωτή και η δημόσια υγεία. Η κυρία Σάτου Χάση έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Ματίας ε, για την εξαιρετική δουλειά της. Οι άνοιες και οι Αλτσχάιμερ είναι τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία και οικονομικό. Υπολογίζεται ότι η φροντίδα ασθενών με Αλσχάιμερ κοστίζει ετησίως 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι περισσότερο ε, από ότι η μείωση ε, κατά 30% των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε κόστος. Και επίση υπολογίζεται ότι διπλασιάζεται ο αριθμό των ασθενών κάθε 20 ετία. Αυτό που χρειάζεται είναι πρόληψη και αξιόπιστη διάγνωση, γι' αυτό και περισσότερη έρευνα. Ε, επί παραδείγματι, πώς επηρεάζουν και πώς βλάπτουν τον ευρικό ε, σύστημα χημικές ουσίες και προάγουν άνοιες ε, τύπου Alzheimer. Γι' αυτό, για λόγους Προφύλαξη θα πρέπει να περιοριστούν, να απογορευτούν τέτοιε ουσίε, όπω είναι φυτοφάρμακα κλπ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα ο συνάδελφος Όουσκι. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, επίτροπε, θα ήθελα να πω κάτι για την νόσο Αλτσχάιμερ. Η έκθεση αυτή δεν έχει βέβαια νομοθετικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια νόσο πάρα πολύ σοβαρή ε, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις και οικονομικές και γι' αυτό ε, είναι και μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα εκτός από ιατρικό. Ε, είναι δε συμφασμένο κατά πολύ με τη γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Τώρα, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μπορούμε να ενισχύσουμε την πρόληψη και αυτό σημαίνει και εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της υγείας των ενδιαφερομένων, αλλά επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού, να τις βελτιώσουμε και να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, να βοηθούμε συλλόγους ε, ε, ασθενών και συγγενών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ούσκη. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Φίλιπ Ζουβά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την νόσο Αλτσχάιμερ έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στα εξή δύο σημεία. Πρώτον, η φύλαξη των ε, βαρέως ε, νοσούντων κατοίκων γνωρίζουμε για λόγους ιατρικούς ότι δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε απότομα το περιβάλλον. Ε, αυτό μπορεί να επιδεώσει ραγδαία την κατάστασή τους και τα συμπτώματα και την νόσο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να παραμένουν στο οικείο τους περιβάλλον οι ασθενείς όσο γίνεται περισσότερο. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις οικογένειες και εκείνους που τους φροντίζουν να μην τις αφήσουμε στη μοίρα τους. Ε, ένα δεύτερο σημείο αφορά την έρευνα. Γιατί την έρευνα. Διότι η ελπίδα είναι ε, να βρεθεί φάρμακο για την αλτσάιμε Και για να βρεθεί φάρμακο χρειάζεται αποτελεσματική έρευνα. Ακούω εδώ και εκεί να λέγεται ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Ίσως ή αναμφίβολα έστω, το δέχομαι. Αλλά εκτός από τα χρήματα θα πρέπει να δούμε και πώς χρησιμοποιούνται. Και μέχρι σήμερα η έρευνα ήταν αλλα εκτο κατακαιρματισμένη, χωρίς προτεραιότητες. Δεξιά και πω χρησιμοποιουνται και μεχρι σημερα η ερευνα ηταν πολυ κατακαιρματισμενη χωρις προτεραιοτητες δεξια και αριστερα ο κόσμος εργάζεται μόνος του και δεν συνεννοείται. Εκείνο που ασχολείται με τη φυσιολογία του κυτάρου, ο κυταρολόγος θα πρέπει πρέπει να συνεννοείται με το φυσιολόγο και ε, τον άλλον ερευνητή για να συντονίζουν τις προσπάθειές τους. Στα κοινά ερευνητικά προγράμματα που ε, άρχισε το συγκεκριμένο πρόγραμμα επί Γαλλικής Προεδρίας. Θα ήθελα τέλος να πω στους ασθενείς και στις οικογένειες ότι προχωρούν τα πράγματα, ότι δεν είναι μόνοι τους και να έχουν εμπιστοσύνη, δεν είναι πια μόνοι τους. Η κυρία ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδης ηγητές για το έργο τους αυτή την έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για την όσο Αλτσχάιμερ και γνωρίζουμε όμως ότι ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η γύρα του πληθυσμού είναι από τις πιο πιεστικές προκλήσεις για το μέλλον. Γνωρίζουμε ότι η άνοια είναι ένας από τους βασικούς λόγους ε, αναπηρίας και εξάρτησης των ηλικιωμένων μας. Ε, σήμερα κυρίως η σύζυγος, ο σύζυγος ή τα τέκνα επομίζονται τη σκληρή δουλειά της φροντίδας ε, του ασθενούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει τροπολογίες και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί μήπως μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για μια καλύτερη παροχή φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στη χρηματοδότηση της έρευνας για νέα φάρμακα για τη θεραπεία ε, των νόσων, αλλά απλά προληπτικά προληπτικά μέτρα ε, που μπορεί να παίρνει ο καθένα, να αλλάζει τη διατροφή του, να αλλάζει τρόπο ζωή. Φαίνεται η διατροφή να είναι πρωταγωνιστή ε, στην εκδήλωση και στην εξέλιξη τη νόσου. Και θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποιου πόρου ε, στην έρευνα εκεί περισσότερο. Το κόστο των ανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 130 δισεκατομμύρια το 2005 και αφορά 19 εκατομμύρια πολιτών ε, ε, ασθενών και ε, νοσηλευτών. Είναι τρομακτική αυτή η νόσος και χρειάζεται περισσότερα. Ο κύριος Χατζημαρκάκης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ καλή η ανακοίνωση και η έκθεση. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Ντάλι και τη συνάδελφο Μάτια. Ε, Κυρίε και κύριοι, το Αλτσχάιμερ είναι μάστιγα τη εποχή μα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την νόσο Αλτσχάιμερ. Άρα, δηλαδή, έρευνα και πάλι έρευνα. Αυτό είναι το θέμα. Ε, πρέπει να ενώσουμε τις ε, δυνάμεις μας ε, και γι' αυτό χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Κομισιόν που είναι να υπάρχει μια εταιρική σχέση, μια καινοτομία για τη γύρανση και για το Alzheimer το, ο καρκίνος ε, παλαιότερα και αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα επίγον. Ε, βέβαια δεν αντιμετωπίστηκε οριστικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες για τον καρκίνο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο Alzheimer. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε προληπτικά, τι θα γίνει στο μέλλον. και ως εκ τούτου, όσον αφορά την πολιτική έρευνα, πρέπει να πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στοχευμένα. Νόσος Alzheimer θα μπορούσε να γίνει ένα θέμα πολύ μεγάλης σημασία. Επόμενη ομιλητρία. Η κυρία Μπρέπολ, σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω αντιπρόεδρο ε, τη Συμμαχία κατά του Αλτσχάιμερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλωσορίζω θερμότατα και ολόψυχα την έκθεση κυρία Ματία. Συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Θα ήθελα όμω το σύντομο χρόνο που έχω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, τη σημασία τη πρόληψη και τη έγκαιρη διάγνωση εκστρατείες συνειδητοποίησης ε, για τα πρώτα συμπτώματα είναι ουσιαστικότατη σημασία, έτσι ώστε και ο ασθενή και ο νοσηλευτή, το συντομότερο ε, και πολύ νωρί να προσφεύγει στη θεραπεία που υπάρχει σήμερα. Και επίσης ε, κοινή κοινοτική έρευνα και ερευνητικά προγράμματα από το 85% της δημόσιας έρευνας Σήμερα δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός συντονισμός και αυτό μοιραία οδηγεί σε επικαλύψεις, σε διπλές ε, ε, έρευνες, σε παράλληλες έρευνες και σε κατακαιρματισμό. Χρειάζεται βελτίωση και της έρευνας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα την αιτιολογία της νόσου και τη θεραπεία της και τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μία για το Catch δεν πρόκειται να δώσω το λόγο σε πάνω από πέντε ομιλητές, να το έχετε υπόψη Ο κύριος Μικολάσικ. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Όσο Αλσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιες βελτιώνει τη μέχρι τώρα κατακαιρματισμένη προσέγγιση που είχαμε στη θεραπεία αυτών των νόσων. Επίσης, ε, με την ανακοίνωση βελτιώνονται οι κοινωνικές συνθήκες για όλο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που οφείλονται και στη ραγδαία γύραση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Στην έκθεση γίνεται λόγος για την ανάγκη επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των νοσηλευτών αλλά και βοήθειας των μελών της οικογένειας. Κάθε χρόνο 1,4 εκατομμύρια περιπτώσεις ε, άνοιας διαπιστώνουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έγκαιρη διάγνωση αλλά και έμφαση στην πρόληψη. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εξασφάλιση της αξιοπρέπειας των ασθενών. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη στην προσέγγιση μας. Επίσης, να μην ξεχνούμε και τα μέλη της οικογένειας των ασθενών, που υπόκειται μερικές φορές σε κοινωνικό στιγματισμό. Η κοινωνία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την προσπάθεια των μελών της οικογένειας που φροντίζουν κατοίκων ε, τους ασθενείς από Αλσχάιμερ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παλέτσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια και τους και εισηγητές, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές ε, άνοιας διαδίδονται με ραγδαίους ρυθμούς. Είτε τα συμπτώματα τα ε, διαπιστώνουμε κατόπιν όταν είναι προχωρημένη η νόσος είτε η θεραπεία δεν είναι επαρκής για τον ασθενή. Θα πρέπει να φέρουμε τις μορφές άγνοιας ως προτεραιότητα της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει επίσης να οργανώσουμε ενημερωτικές εκστρατείες για αφύπνιση του κόσμου ώστε να είναι υποψιασμένο ε, και να εντοπίζει έγκαιρα τα συμπτώματα ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Γιατί επαναλαμβάνω ο αριθμός των ε, νοσούντων από τέτοιες μορφές άνοιας αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Σε πολλά κράτη-μέλη οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών αυτών δεν είναι ικανοποιητικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση και να αναγνωρίσει το, την προσπάθεια των μελών της οικογένειας που φροντίζουν τους ε, ασθενείς στο σπίτι τους. Δυστυχώς ε, δεν μπορώ να σας περιλάβω στο κατάλογο μισό λεπτό μόνο τώρα. Μην ξεχνάτε ότι μιλούμε για Αλτσχάιμερ και γεράσκοντα πληθυσμό, αλλά ε, στην εκλογική μου περιφέρεια είχα έναν 48χρονο ε, που τον φρόντιζε ο πατέρας του, ο ηλικιωμένος πατέρας του, γιατί ο νέος, ο νεότερος, ο γιος ε, έπασχε από Αλτσχάιμερ. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό το θέμα και να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και να μιλούμε βέβαια για συνάφεια της Αλτσχάιμερ με τον γεράσκοντα πληθυσμό, αλλά δεν είναι μόνο πρόβλημα ηλικιωμένων η νόσος Αλτσχάιμερ. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα μιλήσω για την αναφορά. Από το 2007 ασχολούμαι με την περίπτωση αυτή των ε, φθινόπωρο του 2007 έκανα μια ερώτηση προς την Κομισιόν και η ερώτηση ήταν παντελώς ε, ε, ήταν ιδιαίτερα μια ικανοποιητική έκανα λοιπόν συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και με άλλους όλα ήταν ιδιαίτερα σαφή και η απάντηση σας κύριε Ντάλη αυτά που διαβάσατε από εκεί κατέληξα ότι δεν έχετε καμία όρεξη να ασχοληθείτε περισσότερο με το θέμα ε, εσείς όμως ανήκετε σε ένα συλλογικό σώμα σας καλώ λοιπόν και εξ ονόματος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών να μας δώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα ε, με βάση αυτά τα οποία αποφασίστε. Και ε, ε, αν δει κανείς ε, το η συσκευή ε, τότε καταλαβαίνει γιατί κάποιες εταιρείες δεν θέλουν να εμφανιστεί στην αγορά. Αυτό ο σωσπνευστήρας είναι πλαστικός και είναι φτηνός. Όποιος δει λοιπόν πώς λειτουργεί το λόμπι των φαρμακευτικών εταιρεών και όποιος δει ποια είναι τα οικονομικά συμφέροντα για να αποκλειστούν οι μικρές επιχειρήσεις τότε αυτομάτως πολλά καθίστανται αυτονόητα. Σας παρακαλώ λοιπόν σήμερα εδώ να το τοποθετηθείτε με σαφήνεια κατά πόσον θα μα δώσετε τα έγγραφα και κατά πόσον είσαστε πρόθυμο να έρθετε στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να συζητήσετε μαζί μας γιατί οι πολίτες και αυτοί ε, που δεν έχουν αρκετά χρήματα και αυτοί έχουν δικαίωμα μιας σωστή ε, θεραπείας. Πρόεδρο, ε, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και στο πλαίσιο της διαδικασία Catch the Eye θα λάβω πέντε ομιλητέ Λούκα Τσιτσεύσκα, η πρώτη ομιλήτρια κατόπιν μπλικοτσικιούπτε Κάλαχα. Πρώτα κυρία Λουκασεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με το γυράσκοντα πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αύξηση και το αριθμό των νοσούντων από νευροεκφυλιστικές ασθένειε. Τα στατιστικά στοιχεία μα δείχνουν ότι ένα στου πέντε άνω των 80 ετών υποφέρει από την νόσο του Alzheimer, της Βέβαια είναι ανίατη αυτή η νόσο, αλλά με σωστή πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση μπορούμε να επιβραδύνουμε τα αποτελέσματά της. Έχουμε και την ε, έκθεση για το Alzheimer ε, το 2009 και 20% το των νοσούν των παγκοσμίω βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δεύτερη περιοχή μετά την Ασία με τους περισσότερους ασθενείς και στην Πολωνία έχουμε 250.000 ε, νοσούντες από Αλσχάιμερ και μάλιστα υπολογίζεται ότι μέχρι το 2040 θα τριπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Είναι ανησυχητικά αυτά τα στοιχεία γιατί ε, δεν είναι μόνο οι οικονομικές αλλά και οι κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου και δεν πλήττεται μόνο άμεσα ασθενής αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χαίρομαι που το θίγουμε. Μόνο με συνεργασία, με έμφαση στην έρευνα αλλά και με ενημερωτική εκστρατεία μπορούμε να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και να αποτρέψουμε την επέλεση της νόσου. Η κυρία Μπρικεβιτσούτε. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία και τις δράσεις που προτείνεται για την νόσο του Αλτσχάιμερ έτσι ώστε να ε, διασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση, η καλή θεραπεία, η ανταλλαγή κλινικών ε, στοιχείων και ε, επιστημονικής γνώσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα ακριβή στατιστικά στοιχεία για τη διάδοση της Alzheimer. Θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ περιορισμένους δείκτες, πάρα πολύ σαφείς και κλινικά προγράμματα να δώσουμε μεγάλη προσοχή ε, στους επαγγελματίες υγείας και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες που σε καθημερινή βάση ε, φροντίζουν ε, τους ασθενείς. Έγκαιρη διάγνωση, το τονίζω αυτό, χρειάζεται και μια στρατηγική για την πρόληψη της νόσου Αλσχάιμερ με ανταλλαγή στοιχείων και συνειδητοποίηση της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ για την Αλσχάιμερ. Στην Ιρλανδία είναι κάτι που αντιμετωπίζεται που έχουμε ε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, κυρίως οφείλεται αυτό στη γύραση του πληθυσμού ε, και στο μέλλον θα είναι όλο και περισσότεροι ασθενείς. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για την έρευνα, για την αιτιολογία και καλύτερες πρακτικές για τη θεραπεία για την περίθευση. Κυρίως το βάρος αυτό φέρουν οι στενοί συγγενείς. 50.000 είναι εκείνοι στην Ιρλανδία. Και τέλος θα ήθελα να ε, απευθύνω ένα ιδιαίτερο φόρο τιμή στην εταιρεία Alzheimer της Ιρλανδίας που φροντίζει και στέκεται πάρα πολύ στους ασθενείς. Ευχαριστώ κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, απευθύνομαι στον Επίτροπο κύριο Ντάλι. Αυτό το πλαστικό, αυτό που βλέπετε που κρατάς στο χέρι, περί αυτού πρόκειται. Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ε, στη γερμανική περίπτωση είπαν ότι αυτά τα δύο πράγματα ε, συνδυάζονται. Το ένα είναι το φάρμακο και αυτό πρέπει να δοκιμαστεί. Κατ' ουσία πρόκειται εδώ για ένα απλό ε, σωληνάκι. Αν όμως τα βάλει αυτά κανείς τα δύο μαζί, τότε θα προκύψει μεγάλη ζημιά για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη συσκευή μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Είναι λοιπόν σκάνδαλο το ότι η Επιτροπή λέει ότι αυτό το απλό προϊόν θα πρέπει να υποστεί τις ίδιες δοκιμές σαν να ήταν ένα φάρμακο το, ότι το φάρμακο πρέπει να δοκιμαστεί αυτό είναι απόλυτα σαφές αυτό όμως το πλαστικό εξάρτημα ε, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο ε, σημαντικό και δεν μας δόθηκε ικανοποιητική απάντηση. Ε, τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούσαν να αποκομίσουν πολλές εξοικονομήσεις αν επιτρεπόταν να χρησιμοποιείται αυτό το πλαστικό εξάρτημα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι εκφυλιστικές ασθένειες μεταξύ των οποίων και το Alzheimer είναι μια ε, προτεραιότητα υγειονομικής φύσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή εδώ η ασθένεια έχει ε, πολλές ε, σημαντικές συνέπειες όχι μόνο σε επίπεδο αλλά και το υψηλό κόστος για τις θεραπείες άμεσες και έμεσες. Το Alzheimer δεν αφορά μόνο αυτούς που νοσούν αλλά αφορά και όλους εκείνους που ασχολούνται με τους νοσούντες. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα. Ε, συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη, συντονισμένες ενέργειες που αφορούν κυρίως ε, την ε, έρευνα και την επιστήμη. Πρέπει λοιπόν κανείς να ασχοληθεί κυρίως με την πρόληψη και την διάγνωση. Να ασχοληθούμε και με καινοτόμε μεθόδους, να δούμε λιγάκι τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα την ασθένεια. Ε, εντάξει, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάλι έχει το λόγο. Κύριε Πίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο, να τους ευχαριστήσω για τη στράτευσή τους σε αυτή την τόσο σημαντική υπόθεση του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας. Εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου και τις συστάσεις του. Δράτω με τις ευκαιρίες για να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται ε, στο να εξετάσει καλύτερα το Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοια γιατί και αυτές οι δύο ασθένειες εντάσσονται μέσα στη διαδικασία γύρωνσης πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Είναι λοιπόν συλλογική ευθύνη να συνεργαστούμε για να μειώσουμε το βάρος και για να επενδύσουμε στην ε, καινοτομία, ε, στην πρόληψη, στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση των ε, επιπτώσεων. Θα στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια Alzheimer και ε, άλλες μορφές Ε, Τώρα, όσον αφορά την αναφορά του κυρίου Κλάιν, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ε, απευθύνομαι στην κυρία Μαντσόνη ε, που είπε ότι η δουλειά της Επιτροπής είναι να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η δική μου η δουλειά είναι να βρίσκομαι κοντά στους ασθενείς. Για μένα είναι Ω Επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας για μένα είναι πολύ σημαντικό ε, να μην κάνω κανένα συμβασμό όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών να μην ε, περικόπτω τίποτα ούτε να αλλάζω τις ε, διαδικασίες εκείνες ε, που έχουμε για να διασφαλίζουμε ότι οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για ιατρικού σκοπούς οποιαδήποτε λοιπόν συσκευή δοκιμάζεται σωστά και αποδεικνύεται ασφαλής. Εδώ το θέμα που εξετάζουμε δεν είναι το πώς θα χρησιμοποιήσει κανείς ένα φάρμακο από κοινού με ένα πλαστικό εξάρτημα. Το θέμα που τίθεται είναι ότι χρειαζόμαστε κλινικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Και για να γίνει αυτό, ο αναφέρον, σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Κλάιν, εκλήθη να προβεί σε κλινικές μελέτες σε 24 ασθενείς, 24 ασθενείς Αυτά, αυτές είναι οι κλινικές μελέτες που του ζητήσαμε. Γιατί λοιπόν δημιουργείται όλη αυτή η αντίδραση, γιατί διαφωνεί στο να προσφέρει αυτές τις κλινικές μελέτες. Τι του προκαλεί αυτή την αντίδραση και αυτό με απασχολεί και εμένα. Πρέπει το χάρη να γνωρίζουμε ε, αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο φάρμακο, με πολλά είδη φαρμάκων και αν ναι, τότε μήπως απαιτείται και διαφορετική δοσολογία. Υπάρχει δυνατότητα ε, προσαρμογής ε, της συσκευής στη δυσκετική δοσολογία. Εγώ όσα απλός ασθενής, αν επρόκειτο να χρησιμοποιήσω αυτή τη συσκευή, αυτά θα με απασχολούσαν. Και αυτά ρώτησαν ε, και οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν αποδείξεις ότι η συσκευή είναι ασφαλής στα χέρια των ασθενών. Όπως σας είπα λοιπόν προβλέπεται η διαδικασία για τη διασφάλιση της ασφάλειας. Ε, και εγώ δεν μπορώ αυτό ε, να το παραβλέψω πράγματι αναφέρθηκε είχα υποσχεθεί να επιληφθώ της υπόθεση. Το έπραξα. Ασχολήθηκα με αυτήν και ε, μπήκα μάλιστα και σε λεπτομέρειες της υπόθεσης. Προφανώς ε, αυτές οι λεπτομέρειες τις ε, έμαθα από άλλους που βρέθηκαν εδώ στην Επιτροπή από το 1997. Και όταν ο κ. Κλάν ζήτησε να συναντηθεί μαζί μου και με τους συνεργάτες μου, δέχτηκα πάρα αυτά. Να συναντηθούμε, είπα. Ο επικεφαλής, ο διευθυντής του γραφείου μου, του είπε ότι βεβαίως να ε, διοργανώσουμε μία συνάντηση, έστειλε ένα μήνυμα και ανέφερε ε, πάρα πολλές προϋποθέσεις και ως μία προϋπόθεση ε, ανέφερε ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει πλήρως τις δαπάνες, τις δαπάνες του κυρίου Κλάιν και των συνεργατών του. Κάτι το οποίο λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να καλύψουμε αυτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρία Ματίας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα ευγενικά λόγια και την υποστήριξή τους ε, ως προς την έκθεση για την όσο Αλσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική και Γι' αυτό είναι σημαντικό το θέμα της ε, έγκαιρης διάγνωσης. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα ζήτημα που ήταν το κοινό σημείο, κοινός παρανομαστής όλων των παρεμβάσεων. Το θέμα της αξιοπρέπειας των ασθενών, του σεβασμού των δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά όχι μόνο των πασχόντων και των μελών της οικογένειάς τους και των ε, ε, νοσηλευτών ή όσους χωρίς να είναι ειδικευμένοι φροντίζουν ως μέλη της οικογένειας τους πάσχοντες. Χαίρομαι πραγματικά με τα λόγια του Επιτρόπου που είπε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει πολύ θετικά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα κάνει ό,τι μπορεί ο Επίτροπος για να τις θέσει σε εφαρμογή. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι εις βάρος μας, γιατί το θέμα επί και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάρα αυτά. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα και της ψηφοφορίας αύριο, αλλά γνωρίζουμε κύριε Επίτροπε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από μας πολύ περισσότερα από απλή αλληλεγγύη και ηθική συμπαράσταση. Περιμένουν από εμά συγκεκριμένες δράσεις, απτές και κατάλληλες για τα προβλήματά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Δυστυχώ όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσετε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και να μετατρέψετε σε νομοθετική πρωτοβουλία και να εφαρμόσετε και εμπράκτο αυτέ τι συστάσει. Γιατί θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του και να έχουν αξιοπρέπεια και ισότητα. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Ματία. ευχαριστώ όσου έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε, θα ψηφίσουμε αύριο από τις 12. Ήδη έχουμε σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση σε σχέση με το